για να κατανοήσω και εγώ ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του θέματος. Ευχαριστούμε την ε, κυρία Επίτροπο. Τώρα λοιπόν η συζήτηση ε, θα ξεκινήσει με τους εκπροσώπους των ε, πολιτικών ομάδων. Ξεκινάμε με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Τσάιερ.